συζητάμε στα θέματα των ε, ε, ημερησίων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουμε μία ώρα για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της δημοκρατίας και καταρχήν έχουμε το θέμα της Νοτιοαφρικής ε, σφαγή απεργών ανθρακορίχων και η συζήτηση ξεκινά με την κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να